I know that we are competing with Mr. Van Rompuy and Mr. Barroso and uh, who else I don't even know. Φαίνεται πως ανταγωνιζόμαστε τους κυρίους Βαν Rompuy και Βαρόσο και δεν έρχεται κόσμος. Θα αρχίσουμε τη συνεδρίαση υποθέτοντας ότι και άλλοι θα προσέλθουν. Καλωσορίζω όλες και όλους όσοι είστε εδώ για την συζήτηση αυτή για την πολιτική συνοχής Ευρώπη 2020. Θα ακούσουμε τις παρουσιάσεις συμμερασμάτων μελετών που ανατέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. με ευθύνη του Πανεπιστημίου Strathclyde και άλλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενικής Διεύθυνσης Regio. και αυτή θα παρουσιαστεί από αυτούς τους ε, ειδικούς και μετά θα ακούσουμε και τις απόψεις ειδικών που δεν έχουν συμμετάσχει στις μελέτες αυτές. Πρώτα λοιπόν η κυρία Κριστίν Χάμζα για την πρώτη αυτή μελέτη για την ένταξη των εμβληματικών πρωτοβουλειών flagship initiatives στην πολιτική συνοχής. Έχει το λόγο κυρία μου. ευχαριστώ για την πρόσκληση που μας απευθύνατε να προσέλθουμε σήμερα ενώπιόν σας. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω μια μελέτη εντατική και με μεγάλο ε, φορτίο. Αναγκαστικά θα είναι επιφανειακή η παρουσίαση, γιατί έχω μόνο 10 λεπτά, αλλά μετά θα ακούσω ερωτήσεις. Πρώτα, τι κάναμε στη μελέτη μας. Και για να προσελκύσω το ενδιαφέρον σας ώστε να την διαβάσετε ο σκοπός μας, ο στόχος μας ήταν να εξετάσουμε αυτές τις εμβληματικέ πρωτοβουλίες και να εξετάσουμε πώς μπορούν να εφαρμοστούν σε διασύνδεση με τα ταμεία. Πρώτα λοιπόν τις αναλύσαμε, τις ε, εμβληματικές αυτές πρωτοβουλίες flagship initiatives και εξετάσαμε πώς διασυνδέονται με τα ταμεία. Και εκ παραλλήλου κάναμε και μελέτης ε, περιπτώσεων, case studies δηλαδή, των τρεχόντων προγραμμάτων και τη διασύνδεσή του με τι στρατηγικέ τη Λισαβόνα. Στο τέλος της φάσης αυτής της αναλύσεως, καταλήξαμε σε δύο δέσμες συμπερασμάτων. Πρώτα, οδικούς χάρτες για κάθε μια από τις εμβληματικέ πρωτοβουλίε και επίση γενικέ συστάσει για όλα τα επίπεδα που, που, που ε, παρουσιάζουν ενδιαφέρον για αυτές τις ε, πρωτοβουλίες. Αρχίζω με τα συμπεράσματα, διότι νομίζω ότι τα, το βασικότερο ας πούμε, συμπέρασμα από τη μελέτη είναι ότι ο καθορισμός, το earmarking, με θεματικό προσανατολισμό, γίνεται με θεματικό προσανατολισμό και με υψηλή αξία. Αυτό το earmarking και η στρατηγική της Λισαβόνας αποτελούν και την βάση για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και έχουν οδηγήσει σε περισσότερο προσανατολισμό αναθέματα. Δεύτερο, η στρατηγική 2020 ακολουθεί τον δρόμο αυτό σε σωστή κατεύθυνση. Τρίτο, τα ταμεία προσανατολίζονται ήδη στην κατεύθυνση της ε, ε, Ευρώπης 2020. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει κάποια έλλειψη συνοχής ανάμεσα στις διάφορες στρατηγικές και στους διάφορους στόχους και ιδίω τα ταμεία του κοινού στρατηγικού πλαισίου δεν συνδέονται με τις ε, εμβληματικές πρωτοβουλίες. Και υπάρχει και μια έλλειψη προσαρμογής ανάμεσα σε ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές. Αυτό το τελευταίο μελετάτε λόγω και των συμφωνιών και των συμφωνιών ε, εταιρικής σχέσης. Εμείς εδώ γιατί μιλούμε. Μιλούμε για 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στρατηγική Ευρώπη 2020 και βρίσκονται σε διάφορες φάσεις εξελίξεως και σε διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής. Ωστόσο και οι 7 αυτές ε, πρωτοβουλίες έχουν αυτούς τους τρεις στόχους. Ευφυής, διαρκής, βιώσιμη και συμπεριληπτική για τους στόχους δηλαδή του 2020. Η πρώτη μας ανάλυση ήταν αυτές οι εμβληματικές πρωτοβουλίες Πώ διασυνδέονται με τα ταμεία του κοινού στρατηγικού πλαισίου. Εξετάσαμε τους κανονισμούς από τη μια μεριά τον, και του κανονισμού ειδικά των εμβληματικών πρωτοβουλειών από την άλλη μεριά. Είδαμε ότι αυτοί οι κανονισμοί συνδέονται με τα ταμεία EADF και ESF και με το Ταμείο ε, Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο Αλίας. Από την άλλη μεριά η πρόταση κανονισμού για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο δεν συνδέεται με τις εμβληματικές πρωτοβουλίες τόσο εντατικά. Στον κανονισμό ERDF δεν αναφέρονται καθόλου εμβληματικές πρωτοβουλίες. Στο δε κανονισμό ESF υπάρχει αναφορά, γίνεται μάλλον αναφορά σε τρεις εμβληματικές πρωτοβουλίες, Youth on the Move, skills and jobs και φτώχεια. Και από την άλλη μεριά, εξετάζοντας τον πίνακα αυτών, βλέπω ότι οι εμβληματικές πρωτοβουλίες αναφέρονται στα πέντε ταμεία ως τα εργαλεία εκείνα για να υλοποιηθούν οι εμβληματικές πρωτοβουλίες. Εμείς έχουμε βάλει τα διάφορα χρώματα εδώ με την έννοια ότι αυτό το κόκκινο χρώμα λέει ότι είναι, δείχνει ότι είναι έντονα, έντονος ο χαρακτήρας του εργαλείου για την εμβληματική πρωτοβουλία, άρα ειδικότερα, για παράδειγμα, το ERDF αναφέρεται στην ψηφιακή ατζέντα, εφόσον είναι ανοιχτό ροζ το χρώμα, τότε δεν αναφέρεται ρητά, αλλά συνδέεται, συνδέεται με την νεολαία σε κίνηση και μπορεί να υπάρχουν και άλλα εργαλεία για την υλοποίηση της εμβληματικής αυτής πρωτοβουλίας. Και το πολύ πολύ ανοιχτό χρώμα σημαίνει ότι μόνο σιωπηρά παραπέμπει εκεί, δηλαδή δεν αναφέρεται ρητά, ωστόσο έχει κάποια σχέση. Ίσως η διαφάνεια αυτή να σας φαίνεται περίπλοκη. Αυτό που δείχνει ωστόσο είναι ότι οι κανονισμοί των εμβληματικών πρωτοβουλειών αναφέρονται, παραπέμπουν στα πέντε ταμεία ε, του κοινού στρατηγικού πλαισίου από την άλλη μεριά, αυτό δεν συμβαίνει στις προτάσεις κανονισμών των ταμείων ε, του κοινού στρατηγικού πλαισίου. Τώρα, αυτό που κάναμε εμείς τώρα, από όλο αυτό το πακέτο των αναλύσεων, είναι ότι φτιάξαμε πολυδιάστατους οδικούς χάρτες, που απαρτίζονται από τρία επίπεδα, όπου μπορούν να εφαρμοστούν οι εμβληματικέ πρωτοβουλίε. Το πρώτο είναι το ευρωπαϊκό επίπεδο, το δεύτερο είναι το επίπεδο του κράτους μέλους και το τρίτο είναι το περιφερειακό και τοπικό. Η δεύτερη διάσταση είναι το χρονικό πλαίσιο. Σύντομο χρονικό πλαίσιο, τα επόμενα ένα ή δύο χρόνια, μέσο πρόθεσμο, η επόμενη χρηματοδοτική περίοδος και μακροπρόθεσμα είναι πλέον μετά το 2020, πέραν του 2020. Εμείς διακρίνουμε τέσσερις τύπους δράσεων. Πρώτα, τύπος Α, η δράση στρατηγικών, πολιτικών, Β, προγράμματα και εργαλεία, Σ, Γ είναι πιλωτικά προγράμματα, πιλωτικές δράσεις μάλλον και η ευρύτερη εφαρμογή. Εάν βάλει κανείς αυτές τις τρεις διαστάσεις όλες μαζί, μαζί με τον οδικό χάρτη που έχουμε στη μελέτη μας και δεν μπορώ να εξηγήσω βέβαια με λεπτομέρειες τώρα διότι υπάρχει πολύ λίγος χρόνος διαθέσιμος. Πάντως για κάθε μια από τις ε, flagship έχουμε συντάξει τέτοιον οδικό χάρτη όπου μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει κονδύλια από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο σε ποιο επίπεδο, για ποιον τύπο δράσεως και σε ποιο χρονικό πλαίσιο. Σας δείχνω λοιπόν ε, ένα απλοποιημένο μοντέλο που εντοπίζονται οι διαφορές μεταξύ των εμβληματικών πρωτοβουλίων. Για παράδειγμα, Innovation Union. Βλέπετε το μπλε, πολύ σύντομες ε, δράσεις, κόκκινο μέσο πρόθεσμες και πράσινο μακροπρόθεσμες οι στήλες αυτές. Θα δείτε λοιπόν επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, κράτους μέλους και περιφερειακό. Βλέπετε λοιπόν την Innovation Union πολλές δράσεις διαφορετικών τύπων που συγκεντρώνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την άλλη μεριά, skills on jobs, δεξιότητες στην εργασία, ε, είναι κυρίως προσανατολισμένοι στις χώρες μέλη, όπου εκεί μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα στο επίπεδο του κράτους μέλους και ιδίω με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό Βέβαια ποικίλει, αλλά με πολύ απλουστευτικό τρόπο τώρα δείχνει ποια, ποιος είναι ο σχεδιασμός, ποια είναι η σχεδίαση μάλλον των ε, οδικών χαρτών. Εν τέλει έχω τρεις διαφάνειες με περιεχόμενο τις συστάσεις μας. Πάλι κάπως απλοποιημένα. Πρώτα, ε, εάν δημιουργηθούν οδική χάρτες για τις ε, εμβληματικές ε, πρωτοβουλίες, τότε πρέπει να ληφθεί υπόψη η εδαφική συνοχή. Αυτό είναι απαραίτητο, διότι δεν μπορεί να γίνει η Innovation Union με την ίδια ταχύτητα και στο ίδιο βάθος, ας πούμε στις κάτω χώρες ή στην Πολωνία ή στην Ρουμανία. Υπάρχει διαφορά, υπάρχει διαφορά στην εδαφική συνοχή. Μπορώ να βάλω ως παράδειγμα οποιαδήποτε χώρα, δεν εξετάσαμε κάποιες συγκεκριμένες, λέω απλώς ότι υπάρχουν διαφορές αναχώρα και η βάση από την οποία θα αρχίσει κάθε χώρα να εφαρμόζει τις ε, πρωτοβουλίες αυτές. Δεύτερο, η συνοχή μεταξύ ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου και των εμπληματικών πρωτοβουλειών, κατά τη γνώμη μας, δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη. Ή πάντως δεν υπάρχει διασύνδεση και ιδίως στην τρέχουσα πρόταση κανονισμού για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Και τέλος, κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει, τα αποτελέσματα μάθησης, τα learning effects της τρέχουσα τρέχουσας περίοδου δεν χρησιμοποιούνται τα διδάγματα αυτά δηλαδή για τη νέα περίοδο, διότι πάλι μπαίνει νέα ορολογία, νέα συστήματα και δυστυχώ αυτό δεν βοηθάει σε μια καλύτερη εφαρμογή αυτού του πολύ εξελιγμένου, του πολύ περίπλοκου συστήματος αφενός λοιπόν με τη flagship και από την άλλη μετά τα μία του ε, κοινού στρατηγικού πλαισίου. Τώρα, συστάσει ειδικότερα για την εφαρμογή των flagship initiatives για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό προτείνουμε, αλλά βέβαια πρόταση είναι μόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει την ευθυγράμμιση των flagship initiatives και των πολιτικών συνοχών. Στην δε διάρκεια της εφαρμογής των εμβληματικών αυτών πρωτοβουλειών να παρακολουθεί από κοντά την πρόοδο. Για παράδειγμα, με θεματικές ομάδες εργασίας. Όπως είπα, αυτό είναι μια πρόταση απλώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του περιφερειακού και τοπικού επίπεδου. Από αυτό γίνεται ήδη. Και πάλι η τρέχουσα κατάσταση της λειτουργίας του κοινού στρατηγικού πλαισίου άρχισε ήδη να αποδίδει κάποια πράγματα τα οποία δεν γίνονταν όταν εμείς κάναμε τη μελέτη. Αυτό που νομίζουμε όμως είναι ότι στο τοπικό επίπεδο θα πρέπει να υπάρξουν ειδικέ ενδεικτικές συστάσεις για το τι θα γίνει με τις εμβληματικές πρωτοβουλίες. Μπορεί να γίνει ας πούμε αυτό ε, ειδικά με τη χρήση του Περιφερειακού Ταμείου αλλά καθώς και με το ε, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σε άλλο θέμα τώρα, στο επίπεδο δηλαδή των χωρών μελών, θα πρέπει να υπάρξουν συμφωνίες μεταξύ των τοπικών αρχών και των κρατών μελών, διότι συχνά οι αρχές δεν έρχονται σε επαφή αρκετά με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στρατηγικές και τα εργαλεία, τα instrument δηλαδή, γιατί αυτά εκπονούνται εδώ, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Τελευταίο, αλλά σημαντικό, πώς θα μεταφέρουμε τη γνώση Πώ θα μεταφέρουμε την τεχνογνωσία. Το λέω κάθε φορά, αλλά πρέπει να το πω και εδώ, πρέπει να το τονίσω και εδώ. Αυτά και νομίζω ότι σεβάστηκα και το δεκάλεπτο. Αν έχετε ερωτήσεις, επειδή πρέπει να φύγω νωρίτερα, να μου τις υποβάλλετε τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις τώρα από τους συναδέλφου. Όταν φύγετε θα έρθουν, φοβάμαι. Σας ευχαριστώ κυρία Χάμζα. δεν συνηθίζεται να γίνεται αυτό, ε, δεν το συνηθίζουμε, αλλά σήμερα έγινε. Ο Γιάννα έχει μία ερώτηση. Έχω μία φιλοσοφική ερώτηση, κύριε Χάμζα. Όταν διαβάσουμε το κείμενό σας, βλέπω κάτι ενδιαφέρον. Η σχέση με την συνθήκη της ε, Λισαβόνας, μάλλον με τη στρατηγική της Λισαβόνας υπάρχει μια περιπτωσιολογική ανάλυση μετά την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Το φιλοσοφικό ερώτημα είναι το εξής. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ανοικοδομήσουμε τον τρόπο που σκέφτονται οι συντάκτες των εμβληματικών πρωτοβουλειών. Να βρούμε τη λογική τους. Να ξαναβρούμε μάλλον τη λογική που είχαν όταν έγραφαν τις πρωτοβουλίες. Αυτό είναι ένα θετικό συμπέρασμα, ότι δηλαδή σκεφτόντουσαν τα εργαλεία. Δεν νομίζω ότι τα σκεφτόντουσαν. Γράψαν αυτές τις εμβληματικές πρωτοβουλίες, χωρίς να σκεφτούν ε, τα εργαλεία. Και μετά είπαν, να οι εμβληματικές πρωτοβουλίες, εφαρμόστε τις. Εμείς τώρα προσπαθούμε εκ των υστέρων να ανασκευάσουμε, να ψάξουμε να βρούμε τι σκεφτόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι. Πόση σημασία έχει αν πέτυχε ή απέτυχε η Λισαβόνα για τις εμβληματικές πρωτοβουλίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί συχνά λέμε ότι φταίει η μέθοδος, φταίει η μέθοδος της αφήγησης Λισαβόνας, που ήταν η μέθοδος του ανοιχτού συντονισμού που ήταν αποτυχημένος. Αν είναι κακή η μέθοδος, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη μέθοδο ή όχι. Να απαντήσω στο δεύτερο ερώτημα τα συμπεράσματα από αυτές τις περιπτωσιολογικές μελέτες ήταν πολύ ευραία. Το δικό μου συμπέρασμα ήταν ότι καταρχήν τα διαφθορτικά ταμεία χρησιμοποιούνται για πολιτικές των κρατών μελών. Όλοι το ξέρουν, έτσι. Αυτό γίνεται. Σε κάποια κράτη-μέλη αυτές οι στρατηγικές δεν συνδέονται απόλυτα με αυτά που σκέφτεται και κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά βέβαια στην συγκεκριμένη περίοδο προγραμματισμού τα προγράμματα προσαρμόζονται ούτω ώστε να λάβουν υπόψη τι στρατηγικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί λένε. Εντάξει, δεν κινούμαστε προ την στρατηγική τη Λισαβόνα που είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά α προσαρμοστούμε λιγάκι. Στο μεταξύ, ενέσκυψε και η κρίση, όλα ήρθαν τα πάνω κάτω. Ε, έπρεπε να κάνουμε κάποιε προσαρμογέ για να σεβαστούμε κάπω τη στρατηγική τη Λισαβόνα. Το συμπέρασμα είναι ότι η στρατηγική τη Λισαβόνα και η έμφαση σε αυτή τη στρατηγική μας ανάγκασε να επαναπροσανατολίσουμε τη στρατηγική μας και να την κάνουμε πιο ενωσιακή. Αυτό είναι το συμπέρασμα και αυτό είναι πολύτιμο. Γιατί πριν τα εργαλεία αυτά τα, χρησιμοποιούσαμε για όποιες ανάγκες είχαμε. Έτσι, αυτό ήταν το πρώτο. Και το δεύτερο, σε τοπικό επίπεδο, κανένας δεν λογαριάζει τις στρατηγικές Λισαβόνας. Αδιαφορούν πλήρως. και πολλά από τα περίπλοκα στρατηγικά θέματα δεν έχουν γίνει κατανοητά στο τοπικό επίπεδο. Να το πω απλά. Ποιο ήταν το πρόβλημα λοιπόν, ότι μερικές φορές τα κονδύλια μην χρησιμοποιείται, Δεν υπήρξε απορρόφηση των κονδυλίων για κάποια προγράμματα. Και στο τέλος της περίοδου, της περίοδου προγραμματισμού, ε, τα ξοδεύουμε που να είναι τα λεφτά. Αυτό έγινε στην Αυστρία, έτσι. Δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Συνέβη στην Αυστρία αυτό που σας λέω. Τώρα, το, άλλο που είπατε για τους συντάκτες και τη σχέση με τα ταμεία ή τα εργαλεία. Τα, οι προηγούμενες εμβληματικές πρωτοβουλίες δεν ήταν κακές. Οι πρωτοβουλίες αυτέ δεν είναι κακές. Είναι μια βάση. Και σκοπός είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα πιθανά δυνατά εργαλεία για να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Γενικά δεν είναι κακή ιδέα. Α πούμε, η ψηφιακή ατζέντα δεν είναι κακή ιδέα. Υπάρχουν πολλά εργαλεία. Δεν είναι μόνο τα θεία διαρθρωτικά ταμεία. Έχουμε τον ορίζοντα 2020. Η ιδέα ποια είναι να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά και να τα χρησιμοποιήσουμε με συνεκτικότητα. Αυτό το κάνουμε για τι ε, συμφωνίε εταιρική σχέση. Δεν είναι κακή αυτή η ιδέα. Και οι συντάκτε είχαν πει ποια εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν πού. Επίσης, υπάρχει και ο δικός χάρτης. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε έτοιμους οδικούς χάρτες για την αποτελεσματικότητα των πόρων. Τώρα είμαστε στη φάση εφαρμογής των οδικών χαρτών αυτών. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε την ε, χρήση των ε, ταμείων και τη σχέση ανάμεσα στα στους οδικούς χάρτες και στα ταμεία. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια για την έκθεση, θα ήθελα ο κύριος Ματιό Φίχτερ από την Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο να παρουσιάσει τη δεύτερη μελέτη για την έξυπνη εξειδίκευση. Κύριε Φίχτερ. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων που μας δίνει την ευκαιρία να έρθουμε εδώ και να παρουσιάσουμε την εργασία που επιτελέσαμε τους τελευταίους μήνες. Ο στόχος μου μέσα σε αυτά τα 10 λεπτά είναι κάπως σύντομο να σας παρουσιάσω την ε, έκθεση αυτή που αποτελεί και κατευθυντήριες γραμμές για τις διαχειριστικές αρχές. Γι' αυτό λοιπόν θα υπενθυμίσω πρώτα απ' όλα το πλαίσιο της εργασίας ε, που είναι έρευνα και καινοτομία. Στρατηγικές δηλαδή έρευνας ε, και καινοτομία σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό για την ευφύ εξειδίκευση. Έπειτα θα μπω σε λεπτομέρειες όσον αφορά τις συστάσεις που κάνουμε και θα δούμε και τι μπορούμε να περιμένουμε για την νέα προγραμματική περίοδο. Τέλος, θα αναφερθώ σε κάποιες βέλτιστες πρακτικές, γιατί η δουλειά αυτή είναι μια πρακτική δουλειά που βασίζεται σε παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που έχουμε εντοπίσει σε διάφορες περιφέρειες. Πολύ σύντομα, λοιπόν, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη προγραμματική περίοδο έχουμε την εξάντε αιρεσιμότητα όσον αφορά τις στρατηγικές καινοτομίας και έρευνας για την ευφυή εξειδίκευση. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια ευκαιρία να επενδύσουμε στην καινοτομία, αλλά αυτό που μας απασχολεί εμάς και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να δώσουμε την, εξής, ε, την απάντηση στην εξή ερώτηση, δηλαδή πώς μπορεί η περιφέρεια να το πετύχει αυτό στα πλαίσια της νέας πολιτικής συνοχής και πώς μπορεί να επενδύσει και στην καινοτομία και στο περιβάλλον με την εξάντε αιρεσιμότητα. Αυτό είναι και ένας στόχος κλειδί του οδηγού αυτού και της μελλοντική πολιτικής συνοχής. Γιατί υπάρχει αυτός ο οδηγός. Η βασική ιδέα είναι η εξής. Η ευθύς ε, προσέγγιση και η ιδιωσιμότητα είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος που πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Δεν πρέπει να υπάρχει απομονωμένη προσέγγιση και να βάζουμε από τη μια μεριά ας πούμε την καινοτομία και από την άλλη την πράσινη ανάπτυξη. Και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι διαχειριστικές αρχές και να συμπεριλαμβάνουν και τις δύο πτυχές στην ε, στρατηγική τους για την καινοτομία. Θέλουμε να δείξουμε ότι έχει νόημα για τις περιφέρειες να γεφυρώσουν, να δημιουργήσουν συνεργασίες ανάμεσα στην καινοτομία και την βιωσιμότητα, γιατί είναι κάτι θετικό, είναι υπέρ της απασχόλησης και υπέρ της ανάπτυξης. Αυτό το οποίο επίσης βοηθάει πολύ είναι, πρέπει να ξέρετε, πρόκειται για ένα πρακτικό οδηγό. Δηλαδή δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα για περιφέρειες οι οποίες βρίσκονται στο επίπεδο του σχεδιασμού και ετοιμάζουν ε, τα προγράμματά τους. Δίνουμε καλές ιδέες που έχουν ήδη εφαρμοστεί κάπου. Δεν πρόκειται δηλαδή για κάτι εντελώ θεωρητικό. Εμείς ε, το αποδεικνύουμε ότι αυτά που προτείνουμε αποτελούν πραγματικότητα για ορισμένε περιφέρειες. Είναι δηλαδή βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσαν κάλλιστα να αντιγράψουν και άλλε περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιεχόμενο τώρα του οδηγού. Πώς να γεφυρώσουμε λοιπόν αυτές τις δύο πτυχές, την ευφυή προσέγγιση και την βιωσιμότητα. Τι πρέπει να κάνουμε, τι βήματα πρέπει να αναλάβουμε σε περιφερειακό επίπεδο τη στιγμή που σχεδιάζουμε την καινοτομία μας, τις στρατηγικές καινοτομίας πολύ βασικό λοιπόν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αυτό και για όλους επίσης τους ε, εταίρους που ασχολούνται με την καινοτομία. Έχουμε επιλέξει τρία στοιχεία που είναι η οικολογική καινοτομία, τα οικολογικά συστήματα, η βιοοικονομία και η βιώσιμη ενέργεια. Όπως σας έχω ήδη πει, έχουμε 18 βέλτιστες πρακτικές μέσα στον οδηγό αυτό και αναφέρονται για να βοηθήσουμε τις διαχειριστικές αρχές και τους διάφορους φορείς που ασχολούνται με την καινοτομία. Ποια είναι τα μηνύματα κλειδί στον οδηγό αυτό. Πρώτο και κύριο, έχει πραγματικά νόημα να συνδυάσουμε την ευφυή και την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό το δείχνουν και διάφορες κοινωνικο-οικονομικές ε, μελέτες, ότι η καινοτομία οδηγεί σε βιωσιμότητα, αλλά βοηθάει και στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Στους καιρούς αυτούς κρίσης που διανύουμε, δεν είναι πολυτέλεια να γεφυρώσουμε λοιπόν την καινοτομία με την ε, βιωσιμότητα. Πρέπει επίσης να βλέπουμε μακριά συνδυάζοντας ε, τα στοιχεία αυτά μέσα στις στρατηγικές μας για καινοτομία. Όλο και περισσότερο έχουμε στόχο να πάμε σε καινοτομίες που αποτελούν πραγματικές αλλαγές. Είναι αλλαγές τεράστιες που γίνονται στην Ευρώπη και οι περιφέρειες αποτελούν και τον καταλητικό παράγοντα για να γίνουν οι αλλαγές αυτές. Πολύ συχνά βρίσκονται στο κέντρο της ανάπτυξης ή του γεφυρώματος αυτού που λέγαμε πριν, στον τομέα της καινοτομίας και της βιωσιμότητας. Αυτό το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να ψάχνει τις δικές της ευκαιρίες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τονίζουμε κι εμείς. Έτσι κι αλλιώς η προσέγγιση δεν είναι ενιαία και ίδια για όλους. Η κάθε περιφέρεια πρέπει να κοιτάξει, να ψάξει, να βρει τις δικές της ιδιαιτερότητες, τις δικές της δυνατότητες για καινοτομία. Άλλοι μπορεί να αναπτύξει περισσότερο στην βιοοικονομία, για παράδειγμα, την καινοτομία και άλλοι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. με τον οδηγό αυτό εμείς καταλάβαμε ότι όλες οι περιφέρειες, όλοι οι φορείς πρέπει πρώτα να κάνουν μια ανάλυση, να δούνε πού βρίσκονται ακριβώς. Τι δυνατότητες έχουν, τι ικανότητες έχουν και τι αδυναμίες επίσης έχουν, όπως επίσης πού βρίσκονται τα εμπόδια και τι μπορούν να ξεπεράσουν και τι όχι. Γιατί οι περιφέρειες στην Ευρώπη δεν μπορούν να είναι όλες Silicon Valley, εξαρτάται πού βρίσκεται η κάθε περιφέρεια σε ποια ακριβώς είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Γι' αυτό και χρειάζεται πρώτα μια ανάλυση. Επίσης έχει μεγάλη σημασία να δούμε τη ζήτηση και την προσφορά. Το θέμα δεν είναι μόνο να έχουμε ενίσχυση και βοήθεια, είναι να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, πώς να ανταποκριθούμε στις προσφορές που υπάρχουν. Κάτι που είναι επίση πολύ σημαντικό, το είδαμε σε πολλά παραδείγματα, είναι να έχουμε επαφή με πολλούς και διαφορετικού φορείς, να είμαστε ανοιχτοί δηλαδή. Και αυτό το έχουμε διαπιστώσει σε όλες τις βελτιστέ πρακτικές. Η συνεργασία με πανεπιστήμια, με τοπικές περιφερειακές αρχές, μικρομεσαίες επιχειρήσει, εμπορικά επιμελητήρια, οργανισμοί ερευνητικοί. Αν θέλει κανείς ας πούμε καινοτομία στην έρευνα, εννοείται ότι πρέπει να συμπεριλάβει και ενεργειακούς οργανισμούς. Αν θέλει καινοτομία στη δασοκομεία ή στη οικονομία, πρέπει να αναζητήσει τους αντίστοιχους φορείς ως εταίρους. Να λοιπόν, τι μπορεί να κάνει κανείς. Πρώτα απ' όλα για την οικοκαινοτομία. Αυτό έχει να κάνει με την ε, επάρκεια πόρων στην Ευρώπη και την ανάπτυξη της κυκλικής καινοτομίας. Εδώ η καινοτομία έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό είναι η οικοκαινοτομία να εισάγεται σε όλους τους τομείς, γιατί δεν πρόκειται μόνο για τις τεχνολογίες εχμής, πρέπει να τη συμπεριλάβουμε ακόμα και στον τομέα των ε, τροφίμων, σε όλους τους τομείς δηλαδή. Πιο σημαντικό ακόμα είναι ότι διασυνοριακά ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και των περιφερειών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε αυτή την περίοδο κρίσης που διανύουμε είναι πολύ σημαντικό γιατί προσφέρει επιπλέον ευκαιρίες για τους ε, φορείς. Τώρα για τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων. Και εδώ βλέπουμε τι πρακτικές υπάρχουν ήδη που αποδίδουν. Γιατί η φύση δεν αποτελεί μια πολυτέλεια, είναι όμως ένα κεφάλαιο για το μέλλον. Πολλές περιφέρειες σε πολλές χώρες μέλη έχουν αναπτύξει πολύ φιλόδοξες προσεγγίσεις για την βιοοικονομία όσον αφορά τα βιοκαύσιμα για παράδειγμα κλπ είναι μία από τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας στην Ευρώπη, οι κλιματικές αλλαγές, η έλλειψη πόρων, η, τα απόβλητα και ανακύκλωση. Εδώ εμείς υπογραμμίζουμε ότι η βιοοικονομία μπορεί να προσφέρει πολλά, γιατί πολλές περιοχές στην Ήπεθρο έχουν τεράστιο δυναμικό για να ε, προχωρήσουν με δύο προϊόντα και να αποτελέσει αυτό ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, Γνωρίζουμε στην Ευρώπη ότι έχουμε τους στόχους για το 2020. Αν όμως θέλουμε να πετύχουμε κάποιους στόχους για το 2050, η καινοτομία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύουμε ότι πολλές από τις περιφέρειες πρέπει να κάνουν πρώτα την αξιολόγησή τους, δηλαδή να, δούμε, να δούνε πού βρίσκονται, τι ικανότητες έχουν όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Οπότε οι επενδύσεις που θα κάνουν να πάνε σε προγράμματα που να έχουν νόημα, όχι μόνο τεχνικά, τεχνολογικά, αλλά και οικονομικά και κοινωνικά, να είναι βιώσιμη δηλαδή η επένδυση αυτή που θα κάνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα στρατηγικό σχέδιο ε, για την ενέργεια με την οποία μπορεί να βοηθήσει τις περιφέρειες να δουν από πού μπορούν να έχουν χρηματοδότηση. Εδώ βέβαια κάνουμε μια διάκριση στον οδηγό μας. Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε επενδύσεις mainstream που ήδη υπάρχουν και πάνε στις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση που χρειάζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και να διακρίνουμε αυτές τις επενδύσεις με τις καινοτόμες επενδύσεις που πάνε στην καινοτομία, που δείχνουν νέους δρόμους, είτε πρόκειται για συνεργασίες σχημάτων, τα κλάστερς, είτε για οτιδήποτε άλλο. Τέλος, να, κάποια παραδείγματα καλών πρακτικών. Ε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα που μάλιστα βραβεύθηκε φέτος. Είναι από την Αυστρία. Είναι ένα σχηματισμός που έχει να κάνει με καθαρές τεχνολογίες στην περιοχή της Στήρια έχουν επενδύσει τα τελευταία 7-8 χρόνια για να αναπτύξουν ένα σχήμα ευρωπαϊκό για τεχνολογίες όσον αφορά το περιβάλλον και την καινοτομία. Συμμετέχουν όλοι οι φορείς της περιφέρειας, 180 είναι συνολικά που συμμετέχουν στο σχήμα αυτό, είναι εντυπωσιακό ο αριθμός και προσφέρουν επίσης υπηρεσίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τις βοηθούν δηλαδή για να τα πάνε καλά στις δραστηριότητές τους. Έχουν πετύχει πολύ καλά αποτελέσματα γιατί διπλασίασαν τον αριθμό των επιχειρήσεων στην περιφέρεια αυτή. Έχουν δημιουργήσει πάνω από 5.000 νέες θέσεις απασχόλησης και η οικονομική ανάπτυξη είναι τεράστια. Έχει σημασία επίσης να υπογραμμίσουμε την αυτοχρηματοδότησή τους, ενώ ξεκίνησαν με επιδοτήσεις και σχεδόν μηδενικό κεφάλαιο από τους ίδιους, τώρα έχουν ένα 50% περίπου ε, χρηματοδότηση από τους ίδιους. Δηλαδή όχι μόνο προσφέρουν ανάπτυξη και απασχόληση, αλλά έχουν δημιουργήσει και ένα οικονομικά βιώσιμο περιβάλλον. Ο οδηγός υπάρχει στην ε, πλατφόρμα S3. Βλέπετε εδώ την ε, ηλεκτρονική διεύθυνση. Είναι μία από τις πρώτες προσπάθειες ε, πάντως που γίνεται μέσω Υπουργείων, μέσω Υπηρεσιών να συνδέσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις που γνωρίζουμε και έχουν πάει καλά υπέρ της εθιούς στρατηγικής. Ευχαριστώ. υπάρχουν σχόλια ή ερωτήσεις. Μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε για το εξής. Ξέρουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο βοηθάει τις περιφέρειες να προετοιμαστούν για το μέλλον, ειδικά στον τομέα της έξυπνης ε, εξειδίκευσης. Οι περιφέρειες ενδιαφέρονται γι' αυτό. Πώς ετοιμάζονται για το μέλλον ιδρύσαμε αυτή την πλατφόρμα για την περιφερειακή καινοτομία και τις σχετικές στρατηγικές με πάνω από 100 ε, περιφέρειες. Έχουμε μια προσπάθεια αξιολόγηση από ομοτήμων. Δουλεύουμε με τις περιφέρειες τις ίδιες, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουν αυτό το χρόνο και να προετοιμαστούν ούτως ώστε όταν υποβάλλουν αυτές τις στρατηγικές, είτε εθνικές είναι είτε περιφερειακές, να είναι και ποιοτικέ, να είναι καλοσχεδιασμένες, ούτως ώστε να δίνουν τα αποτελέσματα και μέσω της πολιτικής συνοχής. Εμείς ε, γι' αυτό εκδίδουμε και τέτοια έγγραφα. Έχουμε, ας πούμε, οδηγούς για πανεπιστήμια έχουμε για την ευρυζωνικότητα οδηγούς, έχουμε και τέτοιους οδηγούς. Ξέρουμε ότι είναι περίπλοκα τα πράγματα και πολλές περιφέρειες ξεκινάνε από το μηδέν σε αυτόν τον τομέα. Γι' αυτό έχουμε λοιπόν αυτά τα εργαλεία να τους κατευθύνουν, να τους βοηθήσουν να κάνουν ποιοτικό προγραμματισμό. Επίσης κάνουμε και διάφορες εκδηλώσεις στα κρατημέλη, διασκέψεις, εργαστήρια, αξιολόγηση ομοτήμων. Υπάρχει μια πλειάδα μέσων που προσφέρουμε στα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη βοηθούν και το ένα το άλλο σε αυτήν την προσπάθεια αξιολόγησης από τους ομότιμούς τους, δηλαδή το peer review αυτό το περίφημο. Για το οργανόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης δεν είμαστε πολύ καλά ενημερωμένοι. Ε, μια ερώτηση έχω να κάνω λοιπόν γι' αυτό. Εσείς ασχολείστε με την βιώσιμη ανάπτυξη και είσαστε και επικεφαλής ομάδας. Αυτό όμως δεν αφορά, δεν είναι μόνο η έξυπνη εξειδίκευση, είναι και άλλα πράγματα, έτσι. Υπάρχουν διάφορες ομάδες. Πώς δουλεύετε τελικά για να προωθήσετε την έξυπνη εξειδίκευση. Η έξυπνη εξειδίκευση είναι μια, ένα γενικό πλαίσιο Έχουμε και τη βοήθεια της, του ICPTS στη Σεβίλη, δηλαδή έχουμε και τη βοήθεια από επιστήμονες, πέρα από τα όσα κάνει το τμήμα μου. Έχουμε και αυτούς τους τομεακούς οδηγούς, ας πούμε, για την ευρυζωνικότητα, για τα πανεπιστήμια κτλ. Έχουμε αυτό το γενικό οδηγό επίσης και έχουμε και πιο τομεακούς λεπτομερείς ε, οδηγούς. το θέμα της καινοτομίας είναι γενικό. Πρέπει να ξέρουμε πού θα καινοτομήσουμε, σε ποια κατεύθυνση θα πάμε. Αυτός ο οδηγός ασχολείται με την πράσινη οικονομία. Είναι πολύ εξειδικευμένο. Υπάρχουν άλλοι οδηγοί που ασχολούνται, όπως σας είπαμε, με το πανεπιστήμιο, την ευρυζωνικότητα κτλ. κτλ. Δηλαδή είναι ένα τμήμα ενός οικονομήματος αυτό αυτός ο οδηγό. Κοιτάω το εύρο των δράσεών σας. Υπάρχουν και οι έξυπνε πόλει που είναι ένα άλλο στοιχείο. Ασχολείστε και με τις έξυπνε πόλει. Που είναι, που είναι αρμοδιότητα της Γενικής διεύθυνση Ενέργειας. Καθημερινά συνεργαζόμαστε με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Και όπως λέει και ο οδηγό αυτός, ε, υπάρχουν κάποιε πρωτοβουλίε για τις έξυπνε πόλεις, ε, για την αστική ανάπτυξη με μικρές εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Ε, πρέπει να υπάρχει ένα θετικό πλαίσιο για να καινοτομήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τη χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχή. Έχουμε αυτόν τον οδηγό. Συνδέουμε λοιπόν το έξυπνο και το βιώσιμο, ειδικά για την ανάπτυξη των πόλεων. Δηλαδή έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Ο Βίκτορ Μποστινάρου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία ερώτηση. Σε όλους τους κανονισμούς και στον οριζόντιο κανονισμό και στου ειδικού κανονισμούς για τα ταμεία, Μιλάμε για τη δημιουργία θεσμικού και διοικητικού δυναμικού. Το λέμε με μονομανία. Πώς προκύπτει αυτό από αυτά που μας είπατε, πώς από εκεί θα φτάσουμε σε νέες πολιτικές, σε μια νέα προσέγγιση για μια νέα περιφερειακή πολιτική. Η Γενική Διεύθυνση, Ρέτζι, τι θα μπορέσει να κάνει για τις ίδιες τις περιφέρειες αυτές καθεαυτές, ούτως ώστε να βελτιώσουν την τεχνογνωσία τους, τις γνώσεις τους, και το δυναμικό τους για να μπορούν να εφαρμόζουν νέες περιφερειακές πολιτικές με τον τρόπο που μας περιγράψατε πριν. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Αν όλα αυτά παραμένουν για τους ειδικού, για ένα ιερατείο θα είναι λίγα και για λίγους. Η κυρία Χάμζα, μια και θα φύγει, θέλω να τη ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μια μεγάλη ασυμμετρία, όπως είπατε, ανάμεσα στη, στην παρουσία των ταμείων στις εμβληματικέ πρωτοβουλίες και την απουσία αυτών των πρωτοβουλίων στον κανονισμό για τα ταμεία. Τι προτείνετε εσεί, τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος ε, από την ε, απουσία αυτής της αναφοράς στον κανονισμό. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, αυτή την έλλειψη. Αυτό που μπορεί να βοηθήσει είναι αυτέ οι συμφωνίε εταιρική σχέσης που υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος. Γιατί εκεί τα κράτη-μέλη έχουν το καθήκον να κοιτάξουν πέρα από τα διαρθωτικά ταμεία. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ψάξουν και άλλα θέματα όπως ορίζοντας 2020 κτλ. Ε, επίσης υπάρχει και ο δικός χάρτης για τις εμβληματικές πρωτοβουλίες. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε τον κανονισμό και να αναφέρουμε κάθε εμβληματική πρωτοβουλία σε κάθε κανονισμό. Δεν έχει σημασία αυτό. Στην πραγματικότητα αυτό που έχει σημασία είναι η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων στοιχείων Τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν, όλοι πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα διαρθωτικά ταμεία χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση Ευρώπη 2020. Και οι πρωτοβουλίες αυτές, οι εμβληματικές πρωτοβουλίες, είναι τμήμα της Ευρώπης 2020. Ας ενταχθούν στις συμφωνίες, ας λάβουμε υπόψη μας οδικούς ε, χάρτες και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο πρέπει να τα ψάξει αυτά να δείτε τι, γίνεται με τους οδικούς χάρτες. Σημεριζόμαστε Συμμεριζόμαστε απόλυτα αυτό που είπατε για την ε, τεχνογνωσία, ικανότητες, προσόντα, δεξιότητες. Γι' αυτό ακριβώς φτιάξαμε αυτούς τους αυτόν τον οδηγό και άλλους οδηγούς και έχουμε οργανώσει δεκάδες εκδηλώσεις σε όλες τις ε, πρωτεύουσες της Ευρώπης και σε άλλες χώρες μη πρωτεύουσες, ούτως ώστε να δημιουργηθεί αυτό το δυναμικό, ε, να δημιουργηθεί αυτή η γνώση, αυτή η τεχνογνωσία για τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Όταν λέμε ότι έχουμε 102 πιο συγκεκριμένα περιφέρειες που έχουν εγγραφεί σε αυτήν την πλατφόρμα. Αυτό δεν είναι θεωρία μόνο, είναι και πρακτική δουλειά. Την επόμενη εβδομάδα ε, στο Στρασβούργο θα κάνουμε μία προσπάθεια αξιολόγησης ομοτήμων. 20 περιφέρειες θα συμμετάσχουν, ούτω ώστε να παρουσιάσουν τις, τα σχέδια στρατηγικών για την καινοτομία. Από τον κανονισμό θέλουμε να, να φτάσουμε στις πρακτικές λύσεις. Γιατί όπως σας είπα, τα πράγματα είναι περίπλοκα και νέα και θέλουμε να βοηθήσουμε. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν, οι οργανώσεις που ξέρουν να βοηθήσουν. Γιατί υπάρχει πολλή γνώση, σε πολλά κράτη-μέλη ξέρουν τι να κάνουν, γιατί το έχουν κάνει και στο παρελθόν. Το θέμα είναι να το πούν και στους άλλους, να το μοιραστούν. Ε, να βοηθήσουν και τους άλλους στην Ευρώπη μέχρι, μέσω της πολιτικής συνοχής. Η αντίδραση είναι θετική και όλο και περισσότερες περιφέρειες και φορείς και εμπειρογνώμονες συμμετέχουν. Συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και θα είναι πολύ περισσότεροι στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο του κ. Μάρκου Στρίλη από το δίκτυο Bankwatch για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την Ευρώπη 2020. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσουμε την άποψή μας για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Αυτό το μέσο ε, δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό που αναφέρθηκε στην πρώτη παρουσίαση ανάμεσα στις εμβληματικές πρωτοβουλίες των στόχων του Ευρώπη 2020 και των κανονισμών με σκοπό τα προγράμματα και τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Τρία λεφτά. Καταρχήν προσέξτε με πριν ξεκινήσω την παρουσίασή μου. Θα ήθελα να σας δείξω τον ύμνο μας για την καλύτερη δαπάνη των μελλοντικών κονδυλίων από τα ταμεία. Α, ελπίζω να αρχίσει να παίζει. not, you will have to sing yourself. Ποιος να το τραγουδήσετε εσείς τον ύμνο. It worked when, when we tested it. Εμείς το δοκιμάσαμε και δούλευε πριν. Ευχαριστώ. Τι είδαμε. Όταν ξοδεύουμε καλά τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, να μειώσουμε το κόστος, να αυξήσουμε την ε, αποτελεσματική χρήση των πόρων αλλά σε μικρή κλίμακα. Με βάση τους στόχους Ευρώπη 2020 και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες. Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε από την Κομισιόν, που είναι παράτημα στον κανονισμό κοινών διατάξεων, θα μας δώσει το στρατηγικό αυτό πλαίσιο, θα μας δώσει την κατεύθυνση και την καθοδήγηση, μαζί με τις διατάξεις, του κανονισμού, ούτω ώστε να φτιάξουμε μια σχέση με τους στόχους Ευρώπη 2020 και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες. Τώρα θα ακολουθήσει μια παρουσίαση. Έχουμε τους ε, κλιματικούς 2020 20 που είναι οι πιο προφανείς, οι πιο γνωστοί, οι στόχοι για το Ευρώπη 2020, την Ευρώπη 2020. Θέλουμε όμως και την ε, πρωτοβουλία, να αναφέρω και την πρωτοβουλία για την ε, αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων, ε, για την, ε, επίσης η στρατηγική για τη βιοπικιλότητα, για την, να, σταματήσει η Ευρώπη να έχει απώλεια βιοπικιλότητας μέχρι το 2020. Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει και αυτά να είναι στο στόχαστρό μας. Στο παρελθόν, αλλά και σήμερα οι κανονισμοί και οι στρατηγικές ήταν καλές για τους στόχους ε, Ευρώπη 2020 και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες, αλλά δεν το είχαμε εκμεταλλευτεί αυτό σε μεγάλη κλίμακα. Πιστεύουμε ότι το κοινό στρατηγικό πλαίσιο το σημερινό, όπως τροποποιήθηκε, είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στις ευρωπαϊκές στρατηγικές, τους στόχους και τις πρωτοβουλίες και τα επιχειρησιακά προγράμματα και τη συμφωνία εταιρικής σχέσης. Είναι σημαντικό λοιπόν που μπήκε ως παράτημα στον καονισμό κοινών διατάξεων, ούτως ώστε να είναι έτσι πολύ ορατό και να υπάρχει και αυτή η ρητή συμφωνία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Όλα αυτά είναι καλά λοιπόν και μας δίνουν μια συνεκτικότητα. Μας, δίνουν, μας εξασφαλίζουν ένα συντονισμό των διαφόρων εργαλείων που έχουμε για τις στρατηγικές ε, Ευρώπη 2020 και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες. Ένα, η χρηματοδότηση προφανώς των κλιματικών στόχων είναι προφανής. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η βιώσιμη ανάπτυξη να μπει παντού. Δηλαδή αυτή οι οριζόντια διατάξη του άρθρου 7 και του άρθρου 8 του, κοινού, του κανονισμού κοινωνικών, κοινών διατάξεων να μπουν παντού. Ξέρουμε ότι για πολλές αρχές είναι δύσκολο να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό το πράγμα στην πράξη. Ε, δηλαδή να βάλουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη παντού, σε όλες τις δράσεις. Και ακριβώς για αυτό το κοινό στρατηγικό πλαίσιο μας δίνει πολύ ακριβείς ιδέες ε, προς τα που πρέπει να κινηθούμε με τα προγραμματά μας, με τον προγραμματισμό μας. Και μπορεί να μας οδηγήσει ε, σε σωστό σχεδιασμό των ε, προγραμμάτων και των συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Θα σας αναφέρω εντάχει κάποιους τομείς, παραδείγματος το τομέα των μεταφορών. Έχουμε αυτό το κοινό στατικό πλαίσιο που προβλέπει ιεράρχηση και κατάταξη των, προγρα... των έργων για τις μεταφορές ανάλογα με τη συνεισφορά τους που έχουν στην κινητικότητα, στη βιωσιμότητα και στη μείωση βεβαίως των αερίων του θερμοκηπίου. Πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης η σχέση με, το... με τη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές και με το στόχο τη μείωση ε, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά 60% είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε επενδύσει, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα την ανάγκη για μεγαλύτερη κινητικότητα στην Ευρώπη από του ανθρώπου, παράλληλα με τη μείωση των ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αύξηση αυτή τη κινητικότητα των ανθρώπων. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του κοινού στρατηγικού πλαισίου κάτι που αναφέρθηκε και πριν, είναι ότι η βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να είναι πιο απτή όταν επιλέγουμε τα προγράμματα, όταν σχεδιάζουμε τα επιχειρησιακά προγράμματα. Θα πρέπει να επιλέγουμε την πιο συμφερτική λύση που υπάρχει στην αγορά σημαντικό αυτό για να εξασφαλίσουμε τη συνέπεια, να αποφύγουμε επενδύσεις που έχουν αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον, στο κλίμα, για να είναι αποτελεσματικά για, την, για τους πόρους. Επίσης να λάβουμε υπόψη μας και το κόστος του κύκλου ζωής όταν προωθούμε κάποια έργα. Και σημαντικό να προωθήσουμε τις ε, πράσινες δημόσιες προμήθειες. Εδώ το δημόσιο μπορεί να, μας, να είναι ένα όχημα που θα μας εξασφαλίσει μεγαλύτερη και καλύτερη χρήση, αποτελεσματικότητα αν θέλετε χρήση των πόρων. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Πρέπει να ιεραρχήσουμε τα απόβλητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι τμήμα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να ξοδεύονται αναλόγως με την ιεράρχηση, δηλαδή με βάση την ιεράρχηση αυτή των αποβλήτων. Για την μείωση, αποφυγή των αποβλήτων, την ανακύκλωση των αποβλήτων, για το μετριασμό του, της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή σε αυτή την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ο στόχος του 20% του, του ενωσιακού προϋπολογισμού που θα πρέπει να πάει για την, το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και θα πρέπει να εξοδευτεί σε κλιματικές δράσεις. Αυτό θα γίνει πιο ορατό στο μέλλον. Και τελευταίο και σημαντικό, υπάρχουν κάποιες βασικές δράσεις που προτείνει η Κομισιόν. Αυτός ο κατάλληλος που ακολουθεί δεν είναι εξαντλητικός, δεν είναι πλήρης, αλλά δίνει μια καλή ιδέα ε, προς τα που θα κινηθούν τα μελλοντικά προγράμματα και οι συμφωνίε εταιρική σχέση. Το συμπέρασμα ποιο είναι. Έχουμε κάποια εμπειρία για τα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα πρέπει να προωθούν έργα και προγράμματα ε, που να υλοποιούν τους στόχους Ευρώπη 2020. Και το κοινό στρατηγικό πλαίσιο μπορεί να είναι σημαντικό εργαλείο, ούτως ώστε τα κράτη-μέλη, οι διαχειριστικές αρχές να έχουν μια καθοδήγηση για το πώς τα προγράμματα εταιρική σχέσης μπορούν να διαμορφωθούν, ούτως ώστε όλα να είναι συνεπείς με τους ευρωπαϊκούς στόχους. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you. I would like... Ευχαριστούμε πολύ. Ερωτήσεις, σχόλια. Όχι, εγώ να σας ρωτήσω τότε κάτι. Στον κανονισμό έχουμε αυτές τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης και πολλές φορές χρησιμοποιείται η έννοια της εταιρική συμφωνίας. Δεν έχουμε αποφασίσει τελικά πώς θα το ονομάσουμε ακριβώς. Εσείς γιατί μιλάτε για συμφωνίες και όχι για συμβάσεις. Αισθάνεστε ότι είναι καλύτερα έτσι. Δεν είναι κριτική αυτό που κάνω. Απλώς επειδή εμεί ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος να το διατυπώσουμε, γι' αυτό σας ρωτάω. Γιατί εσείς προτιμάτε το ένα από το άλλο. Θα δούμε πού θα καταλήξουμε τελικά, ποια θα είναι η σχέση ανάμεσα των κυβερνώντων και της, των εταίρων. Γιατί μιλάτε λοιπόν εσείς για συμφωνία και όχι για συμβάσεις. Ζητώ συγγνώμη. Βασικά προσπαθούσα να προσαρμοστώ στο λεξιλόγιο του Συμβουλίου, αλλά πράγματι οι συμβάσεις εταιρικής σχέσης πρέπει να έχουν βάρος, δηλαδή μια ποιότητα η οποία να ξεπερνάει τα εθνικά στρατηγικά προγράμματα. Πρέπει να αποτελούν μια κατευθυντήρια γραμμή και πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία για την απόδοση βάσει των στόχων που θέλουμε να επιτευχθούν. Ίσως και τα οικονομικά στοιχεία. Μια που με ρωτάτε λοιπόν να διορθώσω τον εαυτό μου και να πω ότι προτιμάω θα ήταν καλύτερα αν είχα μιλήσει για συμβάσει. Μα εσείς ε, μου λέτε τελικά συμβάσεις, ενώ εμείς λέγαμε πως είναι καλύτερα να μιλάμε για συμφωνίες. Σε πάση περιπτώσει. Εσείς εκπροσωπείτε ένα από, ένα από τους οργανισμούς αυτούς που θα συμμετέχουν σε αυτές τις συμβάσεις, συμφωνίες, εταιρική σχέση στο μέλλον. Ρωτάω λοιπόν εσείς πώς αξιολογείτε την ετοιμότητα, την ε, θεσμική ικανότητα, ιδιαίτερα για τα νέα θα μπορούν από εκεί οργανώσεις να αποτελέσουν πραγματικούς εταίρους. Πιστεύετε ότι είναι έτοιμοι ή ότι πρέπει να βοηθήσουμε εμείς ακόμα για να φτάσουν στα επίπεδα αυτά ικανότητας να μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα και να αναλάβουν και ευθύνες. Οι συναδελφοί μου συμμετέχουν στη διαδικασία του προγραμματισμού που έχει διαρχίσει. Υπάρχουν και οι διάφορες ε, ομάδες εργασίας στις χώρες μέλη το, για τα επιχειρησιακά σχέδια. Το ερώτημα τώρα της ευθύνης και ικανότητας των μη κυβερνητικών οργανισμών έχει δύο πλευρές. Αφενός βλέπουμε ακόμη κάποια εμπόδια για την είσοδό τους με παραγωγικό τρόπο στην διαδικασία προγραμματισμού. Από την άλλη μεριά, σε κάποιο, σημείο, σε κάποιο χρονικό σημείο, βλέπουμε τώρα στην τρέχουσα περίοδο και στις monitoring committees, ότι υπάρχει και πολύ υλικό που πρέπει να επεξεργαστούν. Και ναι, μεν οι συνάδελφοί μου δουλεύουν ήδη εδώ και 17 χρόνια, αλλά είναι και προσωπικές επαφές με τους μη κρατικού οργανισμούς και όπως είπα είναι αυτές οι δύο πτυχές που, τα, που είναι λίγο διαφορετικές. Ό,τι αφορά την ευθύνη, νομίζω ότι σε κάποια στιγμή οι μη κρατικοί οργανισμοί θεωρούνται από ορισμένου ως ταραχοποιοί. Δεν νομίζω ότι είναι αλήθεια βέβαια αυτό ούτε άλλωστε είναι και επιθυμητό. Αυτό που έχουν κάνει οι οργανώσεις μου τους τελευταίους μήνες είναι να εργαστούν στο πεδίο όπως λέμε για να συγκεντρώσουν στοιχεία, για να συγκεντρώσουν τα στοιχεία για τους εθνικούς στόχους, για τις χρηματοδοτικές ανάγκες, τους διαφόρους τομείς, να φτιάξουν δείκτες. Επομένως, η διασύνδεση με το πεδίο, με τις τοπικές κοινότητες, με εκεί όπου πραγματικά ε, χρειάζεται και θα εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα, να βρεθούν δηλαδή οι γνώσεις που ενδέχεται να είναι χρήσιμες στην διαδικασία προγραμματισμού, ε, δεδομένου, ότι είναι δυνατή αυτή η ανταλλαγή. Πρόεδρος, αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια ή ερωτήσεις, τότε ας περάσουμε στον επόμενο ομιλητή. Νομίζω ότι ε, έχουμε ένα, έχουμε κοντά μας τον Έσα Χάλμε, περιφερειάρχη της περιοχής Τάμπερε, από τους μεγαλύτερους φίλους της ε, υπόθεσής μας και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα προσπαθήσω να είμαι ρεαλιστής, ας πούμε, στην προσέγγισή μου και να εξετάσω τα πράγματα που κοιτάζουμε εδώ από την περιφερειακή πτυχή, από την αυτό, από τη σκοπιά αυτών δηλαδή, που παίζουν το παιχνίδι στην ίδια την περιφέρεια. Η περιφέρειά μου έχει περίπου 500 εκατομμύρια κατοίκους. Είμαστε πολύ προσανατολισμένοι στην έρευνα και ανάπτυξη. Διαθέτουμε το 6,6% του ΑΕΠ μας σε ε, αυτή την υπόθεση και πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ε, τις άλλες περιφέρειες. Κάνουμε προσπάθεια δηλαδή να βρούμε τη νέα ιστορία επιτυχίας στην περιφέρειά μας. Ο πατέρας μου μου είχε πει εδώ και δεκαετίες βέβαια ότι ο καλός σχεδιασμός πολύ συχνά ανατρέπεται. Και τώρα αυτό ακριβώς κάνουμε. Για το 2020 βλέπουμε αυτές τις flagships και τις προτάσεις κανονισμού που έχουν προχωρήσει τόσο πολύ. Είναι ο καλύτερος στόχος από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι κάτι που μας ικανοποιεί. Έχουμε λοιπόν καλό σχέδιο. Ε, πρέπει να το φτιάξουμε ακόμα καλύτερο ώστε να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Βέβαια, καμιά φορά, όπως λένε, ο διάβολος κρύβεται στη λεπτομέρεια. Και Πρέπει αυτό να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Πώς αλλάζεται η διαφάνεια. Εδώ, ωραία. Πρώτα λοιπόν, όλα γίνονται κάπου. Και αυτό σημαίνει ότι είτε είναι δημόσιος φορέας στην πανεπιστήμιο, είτε είναι ιδιωτική εταιρεία, όλοι, όλοι διαδικτυώνονται κάπου στον κόσμο. Οι περισσότερες όμως από τις νέες ιδέες προσεγγίζουν οι μεν δε μέσα από τα δίκτυα αυτά. Και ο τρόπος με τον οποίο εμείς προσεγγίζουμε την χρηματοδότηση είναι πώς μπορούμε να φτιάξουμε το στόχο έτσι ώστε να εντάσσεται στους στόχους του 2020, ταυτόχρονα όμως να είναι και προσιτός για τους ε, φορείς στην περιφέρεια. Πρέπει λοιπόν όσο καθαρότερος είναι ο στόχος, τόσο πιο εύκαμπτα να είναι τα μέσα. Να εξηγήσω. Στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, παρόλο που ο προπολογισμό δεν έχει ακόμα εγκριθεί, φαίνεται να είναι τεράστιος, αλλά στο περιφερειακό επίπεδο, εν τέλει σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές προς την κατεύθυνση του στόχου, με αυτά που προσπαθεί να επιτύχει σε αιτήσια βάση ε, ο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Εν τέλει και την περιφέρειά μα το ποσό έρχεται σε λίγα εκατομμύρια. Είναι μικρές οι αλλαγές που μπορεί να προκύψουν δηλαδή ε, για τις πολιτικές. Γι' αυτό ο περιφερειακός φορέας, ο παίκτη δηλαδή, ξεκινά κάνοντας πρώτα μία ερμηνεία των εγγράφων. Δεν μπορούμε να τα δούμε όλα κοιτάμε ποια είναι αυτά τα οποία ταιριάζουν καλύτερα ή, αν το πω ανάποδα, ποια μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα την επίτευξη των στόχων. Και μετά προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειες των φορέων που θα προκαλέσουν τις αλλαγές αυτές. Να δώσουμε δηλαδή υποστήριξη σε κάποιον, αλλά όχι μόνο. Να συγχρηματοδοτήσουμε, να συμμετάσχουμε στις αγορές αυτών των όσων θα μας χρειαστούν. Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε τις ευκαιρίες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της υπερβολικής ρύθμισης. Αν δηλαδή πάρετε την ευκαιρία και την επίλυση του προβλήματος, το πρόβλημα γνωρίζετε που επιλύεται, αλλά για την ευκαιρία μόνο να μαντέψετε μπορείτε αν πηγαίνετε σωστά και όταν έχετε πολύ αυστηρές τυπολατρικές ρυθμίσεις είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί κάποια ευκαμψία για την επίτευξη λύσεων. Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά που προσπαθεί να πετύχει η οργάνωσή μας Innovation Direct, δηλαδή πώς θα φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο θα, ε, με στη βάση του οποίου θα, εξεταστεί εάν είναι σωστός ο δρόμος που προσπαθούμε να κινηθούμε. Αυτό ήδη συζητήσαμε σήμερα σχετικά με τις ε, εθνικές πολιτικές και τις περιφερειακές πολιτικές. Εμείς βλέπουμε συνεχώς τις εθνικές πολιτικές να είναι πιο παραδοσιακές και συντηρητικές από τις πρωτοβουλίες που προκύπτουν από τις περιφέρειες. Και αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη σας για τις συμφωνίες συνεργασίας ή τέλος πάντων συμβάσεις συνεργασίας θέλετε, όπως θέλετε πέστε Αλλά πρέπει να υπάρχουν κανόνες για να προχωρήσουμε. Και νομίζω ότι ο κύριος Φίχτερ είπε προηγουμένως ότι αυτό που είναι σημαντικό στην πολιτική καινοτομία δεν είναι μονάχα η υψηλή τεχνολογία και ο προσανατολισμός προς την τεχνολογία, αλλά μπορούν και χαμηλής τεχνολογίας προϊόντα και υπηρεσίες να γίνουν με τρόπο που αρμόζει στη υψηλή τεχνολογία και να αλλάξουν επομένω δομέ. Όταν προσπαθεί, όταν αναζητεί κανεί νέου δρόμου για την ανάπτυξη. την προπαρασκευή του προγραμματισμού, αυτό που βάλαμε εμείς πρώτο είναι η πραγματική μέτρηση για το τι πετυχαίνει η Ευρώπη το 2020 είναι μπορεί να διεισδύσει η Ευρώπη στις αγορές όπου δεν έχει ακόμα ισχυρή παρουσία. Και αυτό είναι που βλέπουμε και στην περιφερειακή κλίμακα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους της Ένωσης για να στηρίξουμε εταιρείε και πανεπιστήμια μας για να, να προχωρήσουν με επιτυχία στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, να γίνουν οι αλλαγές με τρόπο που να τους επιτρέψουν τελικά να επιζούν, να επιβιώσουν χωρίς υποστήριξη. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι αρκετό μόνο να δαπανώνται σωστά τα χρήματα. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και τους κανόνες. Χρειαζόμαστε ακόμη πιο στοχευμένες, πιο ξεκάθαρους στόχους. Το που πάμε ακριβώς δεν το ξέρουμε ακόμη, αλλά η προγραμματικοί στόχοι, η βιωσιμότητα είναι σημαντικά. ο πρωτοπόρος ρόλος στην τεχνολογία, στην καινοτομία επίσης είναι σημαντικός. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ανταγωνισμού. Όχι να ρίχνουμε τους μισθούς για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα. Να πάμε να παίξουμε στις αγορές που είναι εξελιγμένες και να προωθήσουμε εκεί ευφυείς ε, λύσεις. Εμείς θεωρούμε ότι για να πετύχουν κάποιες αλλαγές χρειαζόμαστε καινοτόμα συστήματα. Ένα νέο συστημικό προσανατολισμό. Αυτό που λέω εγώ mailbox policy. Όχι μόνο όμως. Όχι να περιμένεις δηλαδή, την αίτηση να πέσει στο, στην ταχυδρομική σου θηρίδα. Χρειάζεται να ενθαρρύνεις τους παίκτες να συνενώσουν τις προσπάθειές τους έτσι ώστε να προχωρήσουν σε μια συστημική προσέγγιση. Και τέλος έχω, μια, έχω ένα μικρό παράδειγμα δεν μπορείτε να διαβάσετε τόσο καλά. Πάντως τα πρώτα τρία χρόνια στο Health Bio Cluster όπου είναι, συμμετέχουν πολυτεχνία, ε, βιοιατρικές ε, σχολές, επιχειρήσεις κτλ. συνενών τις προσπάθειές τους. Για τα πρώτα τρία χρόνια λοιπόν, χρειάστηκε πρώτα μια τριετία για να ε, εντοπίσουν πού θέλουν να πάνε και τρία χρόνια τα οποία αφιερώθηκαν σε μικρά έργα στην φάση δηλαδή ε, σκοπιμότητας, feasibility phase και όπως ακούσαμε και από προηγούμενους ομιλητές ότι, ότι αυτό απέδωσε και κάποιες επιστημονικές δημοσιεύσεις και ότι μπορέσαν να ανταγωνιστούν με τρία πολύ σημαντικά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες και να τα πάνε πολύ καλά. Αν αξιολογήσετε έστω ένα έργο και να ρωτήσετε ήταν επιτυχία, δεν μπορείτε να πάρετε απάντηση, γιατί όλο το project είναι μια φάση μόνο μέσα στη δημιουργία του συστήματος. Χρειάζεται δηλαδή ανάλυση και αξιολόγηση του ίδιου του συστήματος, έτσι ώστε ε, να είναι μια φάση σε αυτό που προσπαθούμε εν τέλει να επιτύχουμε. Χρειάζεται λοιπόν ανάλυση, αλλά δεν αρκεί για να δούμε ε, εάν είναι επιτυχία το πρόγραμμα. Αυτό ήθελα να σας πω από τη δικιά μας ρεαλιστική σκοπιά των όσων τα εφαρμόζουμε αυτά στην πράξη. Θέλει κανείς να κάνει σχόλια, να κάνει ερωτήσεις. Yes, yes, Maria. Muchas gracias, muchas gracias, Presidenta, y sobre todo... Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση αυτή που πιστεύω ότι είναι τόσο ενδιαφέρουσα για την ε, ανάγκη καινοτομία και δικτύων. Πολύ καιρό βέβαια έχω απομακρυνθεί από τον ακαδημαϊκό κόσμο, τον κόσμο των πανεπιστημίων. Όμως παρόλα αυτά παρακολουθώ τις έρευνες ε, αριστείας που γίνονται από το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης για παράδειγμα, το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο δηλαδή της Μαδρίτης. Και μου αρέσει να ακούω ότι οι ερευνητές μας κάποια στιγμή πάβουν να χρειάζονται ενισχύσεις, κρατικές ενισχύσεις δηλαδή, κονδύλια για να συνεχίζουν την έρευνά τους. Και αυτό το συνδέω και με κάτι που άκουσα πριν από μερικές μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, που έλεγε ότι τρεις ερευνητές Ισπανοί από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο ε, στην Μασαχουσέτη βραβεύτηκαν γιατί έφτιαξαν κάποιο είδου ρομπότ που μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρές ασθένειες. Και αυτό που τραβά την προσοχή μου είναι ότι από τη μια μεριά υπάρχουν λίγα κονδύλια από πλευρά των επιχειρήσεων για να βοηθήσουν τους μικρούς ε, ερευνητές. Από την άλλη, εγώ δεν ξέρω, αυτό το δίκτυο ερευνητών υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν κάποιο πανεπιστήμιο αρχίζει τη διαδικασία με κάποια συγκεκριμένη μελέτη υπάρχει δυνατότητα να συνεχίσει και τα κονδύλια αυτά να χρησιμοποιούνται έτσι πιο αποτελεσματικά. Σήμερα, εξάλλου, που έχουμε δίκτυα, το βλέπουμε αυτό από διάφορες ε, δράσεις, όταν ένας ασθενής είναι σε ένα μέρος και κάποιος άλλος ε, αλλού συνδέονται κάπως οι ειδικοί για την έρευνα. από τους ερευνητές που έχουμε στην Ευρώπη και ξέρω ας από την Ισπανία ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μπορούν όλοι αυτοί να συνδεθούν ώστε σε περίοδο κρίσης όπως είναι η σημερινή να μπορούν να συνδεθούν και έτσι πιο εύκολα να καταλήγουν σε αποτελέσματα για την έρευνά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όπως ε, μπορεί να είδατε και στη διαφάνεια, η οποία ήταν λίγο όμως ε, μικρή, υπάρχει μια σαφής διαφορά ανάμεσα στην υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων από τα διαρθωτικά ταμεία και τα επιστημονικά προγράμματα που προωθούν την έρευνα. Πρέπει να έχουμε τις διάφορες φάσεις για να υπάρξει σωστή χρηματοδότηση. Για το δίκτυο. Αν το πανεπιστήμιό σας λειτουργεί σε αυτούς τους τομείς, σίγουρα έχει επαφές με αυτήν την Ακαδημία όπου υπάρχουν 250 επιστήμονες που συνεργάζονται Πολλά πανεπιστήμια είναι δικτυωμένα. Το βασικό μου μήνυμα είναι ότι να δημιουργήσουμε νέες επαφές πέρα από τις παραδοσιακές, να υποστηρίξουμε τη διαρθρωτική φάση, να βοηθήσουμε τη δημιουργία αυτών των επαφών. Είναι πολύ σημαντικό. Ε, να υποστηρίξουμε τα πανεπιστήμια, η συνεχεία έρχεται και η αγορά και χρηματοδοτεί. Βέβαια, εγώ δεν είμαι βαθύ γνώστη, δεν μπορώ να σχολιάσω το ισπανικό παράδειγμα, αλλά σίγουρα υπάρχουν οι επαφές. Ποιος είναι ο ρόλος των τοπικών αρχών στη δημιουργία αυτού του συστήματο που λέτε, στη δημιουργία αυτή τη δικτύωση. Έχουμε τρεις ρόλους. Πρώτον, να δημιουργήσουμε πλατφόρμες, καταρχήν, ούτως ώστε οι παίκτες που κανονικά δεν συναντούνται, εμείς δημιουργούμε αυτή την πλατφόρμα για να τους φέρουμε σε επαφή. Χρειάζονται λοιπόν και βοήθεια εκτός των πανεπιστημίων, ούτως ώστε τα τα πολυτεχνία, ε, οι ιατρικές σχολές κτλ. να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να βρουν και τα εργαλεία για να έρθουν σε επαφή. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Εν συνεχεία, έχουμε το επίπεδο της περιφέρειας. Ε, η περιφέρεια καλό θα είναι να έχει την παράδοση, να γνωρίζει πώς και να καινοτομεί. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν φορείς στα δημοτικά συμβούλια, περιφερειακά συμβούλια κτλ. που γνωρίζουν τον τρόπο και τη μέθοδο για να βοηθήσουν αυτούς τους φορείς που δεν γνώριζαν αυτή τη διαδικασία έτσι, γονιμοποίησης μέχρι τότε για να τους βοηθήσουν. Και μετά είναι και η φάση η επόμενη, όπου παίρνουμε και ένα ρίσκο, όπου κανένας άλλος δεν πιστεύει ότι αυτός ο τομέας αξίζει τον κόπο να τον προωθήσει. Εκεί έχουμε μια ευελιξία από τους περιφερειακούς φορείς, Αν ας με ρωτήσουμε το κρατικό επίπεδο, τι αξίζει αυτός ο τομέας. Δεν θα μας απαντούσαν καν για αυτή την Ακαδημία. Ε, πού να σκεφτούν τώρα να φέρουν σε επαφή αυτούς τους ανθρώπους, πού να, φέρουν, να πιστέψουν σε αυτή την αλλαγή. Ο ρόλος μας είναι λοιπόν ότι αυτά που απαιτεί η περιφερειακή ανάπτυξη τα προωθούμε. Ε, και τα προωθούμε εμείς γιατί δεν πιστεύουμε ότι ο δημόσιος φορέας είναι ικανός να βρει το κλειδί ας πούμε για αυτή την επιτυχία. Χρειάζεται μια τρέλα. Χρειάζεται έτσι ένα ρίσκο. Να θες να πάρεις ένα ρίσκο για να πετύχεις αυτά τα πράγματα. Η περιφέρεια εκεί μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Ένα νέο ρόλο. Αν κοιτάξετε τα διαφορετικά ταμεία και τον ορίζοντα 2020, τα διαφορετικά ταμεία μπορεί να παίξουν αυτό το ρόλο. Ε, σε αυτή την αρχική, την, την πρωταρχική φάση, ας πούμε, για να φέρουν σε επαφή τους ανθρώπους. Να σας πιέσω λιγάκι. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι όπως πριν δεκαετίες, όπου είχαμε μια χαρά ωραίες ιδέες, πηγαίναμε στον καρά, φτιάχναμε κάτι και μετά έδινε στην αγορά. Δεν είναι έτσι σήμερα. Εσείς είπατε ότι τα προγράμματα, τα έργα τα είναι ένα, μια, ένας κρίκος. Δεν φτιάχνεις πρώτα το σύστημα ε, και μετά λες ποιος θα καινοτομήσει. Γίνεται διαφορετικά σήμερα το πράγμα. Αυτό όμως σημαίνει ότι είναι και πιο δύσκολο, πιο προκλητικό το όλο θέμα. Πρέπει τα καλά προγράμματα, τα καλά έργα, ε, να τα προωθήσεις, ενώ δεν υπάρχει το σύστημα ακόμη ας πούμε, που τα προωθεί από μόνο του. Αυτή την πρόκληση πώς την αντιμετωπίζετε. Έχουμε διάφορα, διάφορες αρένες, πλατφόρμες, πώς να τις πω, καινοτομίας. Όσοι έχουν καινούριε ιδέες, λοιπόν, εκεί μπορούν να τις τεστάρουν. Και στην περιφερειακή ανάπτυξη έχουμε μία πολιτική μια γραμμή πολιτικής, ούτω ώστε να προωθήσουμε αυτές τις πλατφόρμες. Εγώ προειδοποιώ τους δικαικούς μου συνέχεια ότι η πολιτική καινοτομία μια μεγάλη επιχείρηση είναι η τυποποίηση. Γιατί υπάρχει και ο φόβος της μήνυσης. Θα πρέπει να μπορείς να δημιουργήσεις μια πλατφόρμα καινοτομίας, να την προσαρμόσεις στους παίχτες που θέλουν να τεστάρουν τις νέες ιδέες τους. Γι' αυτό η πλατφόρμα αυτή, η αρένα, ο χώρος αυτός πρέπει να είναι ευέλικτος και όλες αυτές οι ανοιχτές πλατφόρμες καινοτομία. είναι ευέλικτες, δεν είναι τυποποιημένες, ευτυχώς, γιατί εκείνη η αξία τους, στη διαφορετικότητά τους. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω περισσότερα για αυτό το θέμα. Αυτή είναι η προσέγγισή μας. Έχουμε και άλλους τομείς όπου αν τους συνδυάσουμε όλους, δημιουργούμε μια ομάδα ειδικών που ψάχνουν να βρουν τρόπο για να καινοτομήσουν στην πλατφόρμα δηλαδή και μετά από την πλατφόρμα φτάσουμε σε ένα μονοπάτι και μετά να χρηματοδοτήσουμε τα πρώτα, τις πρώτες φάσεις του μονοπατιού για να φτιάξουμε μεγαλύτερα προγράμματα εν συνεχεία και να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση ειδική ανάλογα με τον τομέα. Πάμε, τώρα σε μια άλλη περιοχή. Ο Έρικ Μπέσκριτς είναι από την περιοχή αυτή. Παρακαλώ πολύ, από το Bottom. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να έρθω εδώ και να σας πω πώς δουλεύουμε εμείς με την συνοχή και πώς επηρεζόμαστε από την πολιτική συνοχής σε 10 λεπτά, εντάξει θα ξεκινήσω από τα γενικά και θα πάω στα ειδικά μετά. Στον κόσμο βλέπουμε ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους όλο και περισσότερα και ότι όλα συμβαίνουν όλο και πιο γρήγορα. Βλέπουμε επίσης ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε περισσότερο συνδεδεμένοι μεταξύ μας και για μας στη Σουηδία, εντάξει, είμαστε πόσο καιρό μαζί σας, 17 χρόνια που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργαζόμαστε με την Ευρώπη, συνεργαζόμαστε με άλλες περιοχές και συνεργαζόμαστε βέβαια και σε τοπικό επίπεδο. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα και θα σας δείξω πώς μας έχει επηρεάσει εμάς η πολιτική συνοχής και πώς εμείς επηρεάζουμε την πολιτική συνοχής. Όμως, όσα συμβαίνουν, συμβαίνουν σε τοπικό επίπεδο και παίζει ρόλο το από πού προερχόμαστε και πού ζούμε. Εμείς βρισκόμαστε στον, στο βόρειο-βόρειο τμήμα της ε, Ευρώπης. Είμαστε μια περιοχή λίγο μεγαλύτερη από το Βέλγιο. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες αλλά και προβλήματα. Δυνατότητες όμως και ευκαιρίες για να ειδικευόμαστε, να δικευτούμε σε κάτι. Σίγουρα υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ μας. Είμαστε μια περιφέρεια με πλούσιους ε, πόρους, ε, δασοκομεία, ορυκτά, έχουμε χαλκό, χρυσό. Και κυρίως έχουμε ανθρώπινο δυναμικό. 250.000 ε, περίπου άνθρωποι, φοιτητές, ανώτατη εκπαίδευση. Και έχουμε και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας άνεμο, υδροελεκτρική ενέργεια. Τώρα, που οδηγεί η συνοχή, που δεν συζητιούνται μερικές φορές. Είναι κάτι που σιωπηρά το ξέρουμε όλοι, αλλά καλό θα ήταν να το ανακαλύψουμε. Αν συγκρίνουμε πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση πώς έχει κατάσταση, γιατί βέβαια όλα αυτά τα πράγματα θέλουν χρόνο, έτσι δεν πρέπει να είναι κανεί ανυπόμονο, αν θέλει να δει τι επιπτώσει τη συνοχή και τα θετικά. Αν μετά όμω από τόσα χρόνια, αν κοιτάξουμε λίγο πίσω, βλέπουμε ότι είχαμε ευκαιρίε εκμάθηση. Δηλαδή, επειδή είχαμε τα προγράμματα αυτά, επειδή είχαμε την πολιτική συνοχή, είχαμε διαρθρωτικά ταμεία, το κοινωνικό ταμείο, είχαμε πολλές δυνατότητες να συνεργαστούμε και πόρους για να συνεργαστούμε. Αυτό οδήγησε στο να έχουμε και μεγαλύτερες συνεργασίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό από την πολιτική συνοχή, ότι δηλαδή συνεργαζόμαστε περισσότερο σήμερα μεταξύ μας, με τους γειτονές μας, με άλλες χώρες. Οπότε είχαμε ευκαιρίες να μάθουμε από τις συνεργασίες αυτές και να δημιουργήσουμε δίκτυα. Τώρα για περιφέρειες που δεν είναι πυκνοκατοικημένες, αυτό πάντα είναι ένα θέμα. Παρ' αυτά έχουμε φτιάξει αυτό που λέμε την κρίσιμη μάζα, δηλαδή να μπορέσουμε να επωφεληθούμε από τις ευκαιρίες αυτές. Σε συνεργασία με άλλες περιφέρειες στη χώρα μας ή και εκτός. Η οικονομική πόρη τώρα. Όταν είσαστε μια περιφέρεια 600 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα, η οικονομική πόρη είναι πολύ σημαντικό και ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν χρηματοδότηση αλλά και σαν ευκαιρίες για την διάδοση ιδεών, για το πώς μπορούμε να βρούμε πόρους και από όλες τις πηγές επίσης. Όταν διαπιστώνουμε ότι έχουμε κοινά προβλήματα, ε, φτιάχνουμε πλατφόρμες για να τα λύσουμε. Φτιάχνουμε δομές δηλαδή που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές διαφορετικές ε, περιοχές. Και δημιουργούμε και τις κατάλληλες δομές φυσικά για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Δουλεύουμε σε τρία επίπεδα, το μακροπεριφερειακό, το επίπεδο ΝΑΤΣ 2, αλλά επίσης και το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Και έχουμε δημιουργήσει οργανώσεις που κάνουν ακριβώς αυτό. Σε περιφερειακό επίπεδο συνεργαζόμαστε με τις περιφερειακές στρατηγικές και εμβληματικές πρωτοβουλίες οι στόχοι του 2020 είναι πράγματα τα οποία εμείς ήδη δουλεύουμε και εντοπίζουμε παράγοντες για τη δικιά μας ε, ανάπτυξη. Άρα χρησιμοποιούμε σαν δομή του στόχου του 2020. Είναι ήδη η προτεραιότητα για μας. Και σίγουρα θα υπάρχει διαφάνεια για να δούμε αυτό που κάνουμε εμείς και αυτά που γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς συνδέονται. Δουλεύουμε στο δίκτυο NSPA που είναι το δίκτυο για τις λιγότερο κατοικημένες ε, περιφέρειες έχουμε βρει τρόπο να συνεργαστούμε και να εντοπίσουμε λύσεις από τις οποίες να μπορούμε όλοι να υποφεληθούμε. Ε, έτσι βέβαια ενημερωνόμαστε περισσότερο στη Βόρεια Ευρώπη και για το τι ισχύει στην Ευρώπη, αλλά και η υπόλοιπη Ευρώπη ενημερώνεται περισσότερο για το τι συμβαίνει εκεί που είμαστε εμείς. Έχουμε, όπως σας είπα, και μακροπεριφερειακή συνεργασία στην, ε, στην Σουηδία καλύπτει το 50% της, του εδάφους της Σουηδίας, αλλά αφορά μόνο το 10% τον πληθυσμό. Με άλλες αντίστοιχες περιφέρειες λοιπόν βλέπουμε πώς μπορούμε να υποφεληθούμε από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ε, ουσιαστικά ετοιμάζουμε τους αυτούς μας για να συνεργαζόμαστε καλύτερα. Υπάρχει βέβαια και η στρατηγική της Βαλτικής και εκεί συμμετέχουμε. Το επίπεδο ΝΑΤΣ 2 τώρα. Αυτό το επίπεδο είναι επίπεδο διαρθρωτικών ταμείων. Μας έχει δώσει την ευκαιρία να συνεργαστούμε με τους γειτονές μας στην περιοχή και βλέπουμε ότι μπορούμε να αναπτύξουμε πολύ καλύτερα πρωτοβουλίες μαζί τους παρά μόνοι μας όπως κάναμε πριν. Έπειτα έχουμε παραδείγματα και προγράμματα από την συνεργασία αυτή που μας βοήθησε να συμμετέχουμε καλύτερα στη συνοχή. Τώρα υπάρχει κάτι που έχει να κάνει και με τις εμβληματικέ πρωτοβουλίες είναι η επικοινωνία. Αν δεν υπάρχει επικοινωνία για τη δουλειά που κάνεις, δεν μπορείς να επωφεληθείς για καμία από αυτές τις ε, πρωτοβουλίες. Επικοινωνεί επίσης και με τον κόσμο. Αν πάτε στην ψηφιακή ατζέντα θα δείτε ότι εδώ και 10-15 χρόνια πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ έχουν χρησιμοποιηθεί για να αναπτυχθούν δίκτυα στην περιοχή μας και έχουμε τα καλύτερα δυνατό στον τομέα αυτό το ψηφιακό και είναι πολύ βασικό αν θέλει κανείς να ενημερωθεί και για άλλα πράγματα, δεδομένου ότι είμαστε κάπως απομονωμένοι, μακριά από το κέντρο. Μας βοήθησε επίσης η πολιτική συνοχής να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και τις ανάγκες μας ως αεροκατοικημένη περιοχή. Πώς θα αντιμετωπίσουμε ζητήματα υγείας ή άλλα που έχουν να κάνουν με την ευρυζωνικότητα. Συνεπώς, όταν εμείς προβλέπουμε λύσεις ε, ηλεκτρονικής υγείας, ακριβώς επειδή είμαστε μακριά από τα κέντρα, αυτό είναι η ιδιαιτερότητα της δικιάς μας περιοχής. Στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει το αντίθετο. Να υπάρχει μεγάλο ποτηλιάρισμα και αυτό να αποτελεί μια δυσκολία. Να είναι υπερβολικά πύκνο κατοικημένη η περιοχή. Οι εμπειρίες λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Κάποιες ανάγκες μπορεί να τις είδαμε εμείς πρώτοι και να μπορούμε να βοηθήσουμε την Ευρώπη, αλλά βέβαια και αλλιώς και ανάποδα λειτουργεί αυτό. Το θέμα είναι πώς θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Έχουμε φυσικούς πόρους όπως σας είπα, Έχουμε χρησιμοποιήσει ευρωπαϊκά κονδύλια για να τους εκμεταλλευτούμε βιομάζα, για παράδειγμα, για να φτιάξουμε βιοκαύσιμα, ε, βιοαέριο, ε, θέρμανση. Ίσως για την υπόλοιπη Ευρώπη η ψήξη είναι κάτι που χρειάζεται πιο πολύ από την θέρμανση. Εμείς τη χρειαζόμαστε πιο πολύ. Επίσης πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε και τις αδυναμίες. Το ότι δηλαδή έχουμε πάρα πολύ χώρο Όταν ε, η Facebook ήθελε να φτιάξει ένα κέντρο, ήρθε σε εμά επειδή έχουμε χώρο και έχουμε και ενέργεια. Άρα λοιπόν μια δυναμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί θετικά μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη και να αποφεληθεί από αυτή ολόκληρη Ευρώπη. Συνεπώ έχουμε και εμεί δυνατότητε και από τι δικέ μας δυνατότητε μπορούμε να δημιουργήσουμε δυνατότητε και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Είτε για το Facebook όπως σας είπα, είτε αν πρόκειται για άλλου είδου διαστάσεις. Αν κάποιο θέλει για παράδειγμα να δοκιμάσει ένα αυτοκίνητο, μπορεί να πάει στη Βόρεια Φιλανδία και εκεί να μπορέσει να το δοκιμάσει. Μεταπητική βιομηχανία επίσης από τα ορυκτά. Και εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα πληροφορικής που βοηθάει να δημιουργηθούν και νέες θέσεις απασχόλησης. Κάτι το οποίο έχουμε γνωστοποιήσει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί υπάρχουν ίδιες προκλήσεις και τέτοια προβλήματα και αλλού στην Ευρώπη και μερικές φορές και ίδιες δυνατότητες. Έχουμε επίσης ξυλία, δάση. Πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε την ε, ξυλία αυτή. Έτσι κι αλλιώς μπορείς να φτιάξεις και αποθήκες ε, και μάλιστα με ανανεώσιμα υλικά ανακυκλούμενα. Κάτι το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη για να αναπτυχθεί έτσι καλύτερα και η υπόλοιπη Ευρώπη και ο υπόλοιπο κόσμος. Δηλαδή βλέπετε ότι από κάποιες ιδιαιτερότητες μιας περιφέρεια μπορεί κανείς να έχει ιδέε για να αναπτύξει κάποια συστήματα σε άλλες περιοχές και να μπορούν έτσι να αναπτυχθούν παραδέρα και εκείνες. Συνεπώς, όταν οικοδομούμε την Ευρώπη πρέπει και να την οικοδομήσουμε και να την έχουμε έτοιμη, ολόκληρη και συγκροτημένη. Δεν μπορεί να πηγαίνει προς πάσα διαφορετική κατεύθυνση. Τα κονδύλια, η συνεργασία, οι ιδέες από τη συνοχή, η χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων μας, το ότι μαθαίνουμε από άλλους, Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία εμάς μας έδωσαν περισσότερες δυνατότητες για ανάπτυξη και ενισχύουν επίσης και τις δυνατότητες ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αλλά πρέπει να δούμε πόσο δικές μας ιδέες, τα δικά μας ευρήματα, δικές μας επιχειρήσεις και προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υπόλοιπη Ευρώπη για να δημιουργήσουμε ακριβώς μια καλύτερη Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα τους στόχους του 2020, έχουμε δει που βρισκόμαστε σήμερα στην δικιά μας την περιφέρεια και που θέλει η Ευρώπη να πάει. Πιστεύουμε ότι είναι ένα καλό σημείο καμπής, γιατί έτσι ξέρουμε που βρισκόμαστε και μπορούμε να μετρήσουμε και να ξαναμετρήσουμε βάσει των στόχων του 2020. Μπορούμε να αποτελέσουμε ένα παράδειγμα και να συμμετάσχουμε σε όλους τους τομείς για να φτιάξουμε ένα καλύτερο χώρο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τέλος, βλέπουμε ότι τα περισσότερα πράγματα που κάνουμε είναι, έχουν να κάνουν με τις εμβληματικές πρωτοβουλίες και έτσι βλέπουμε και πώς η συνοχή έκανε τη διαφορά σε περιφέρειες όπως είναι η δικιά μας, αλλά και σε, στην περιοχή γενικότερα. Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε την συνοχή στην Ευρώπη, θα έπρεπε να την εφεύρουμε. Σας ευχαριστώ. Thank you very much indeed for your... Ο Προεδρεύων κ. Σταυράκα, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Ποιος από τους συναδέλφους επιθυμεί να λάβει το λόγο. Φαίνεται πως δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν. Και προχωρούμε στο τελευταίο θέμα της ημερησίας διατάξεως μας. Περιφερειακές στρατηγικές για βιομηχανικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Γκάιερ μακρά ημέρα σήμερα και κοπιαστική, γι' αυτό και δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Και εγώ νομίζω ότι είδαμε όλοι ότι από την κρίση μπόρεσαν να βγουν οι χώρες εκείνες μέλη που διαθέτουν μια βιομηχανική παραγωγική βάση. Δείχνει λοιπόν η έκβαση της κρίσης τι μεγάλη σημασία έχει για την ευρωπαϊκή οικονομία και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο η βιομηχανική βάση παραγωγής. Εδώ υπάρχουν δύο στρατηγικές προσεγγίσεις για να διατηρήσουμε. Η μία προσέγγιση είναι οι πρωτοβουλίες βιομηχανικής πολιτικής που προβάλλονται και υποβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελούν στην βάση το ουσιαστικό πλαίσιο. Το εδαφικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο. Η έκθεση πρωτοβουλίας μου θα περιστραφεί γύρω από το πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο να χρησιμοποιηθεί με καλύτερο τρόπο για την διατήρηση και εξέλιξη της βιομηχανίας στις βιομηχανικές περιοχές της Ευρώπης. Βιομηχανική πολιτική από τη μία μεριά, διαρθρωτική αλλαγή από την άλλη. Αυτοί είναι οι δύο πυλώνες στους οποίους θα βασιστεί η ανταγωνιστικότητα των περιφερειών. Με ενδιαφέρει πώς μπορεί η οικονομική βάση, ιδίως στις παλαιές βιομηχανικές περιοχές, να επανεφευρεθεί αν θέλετε ποιες ικανότητες, ποια skills είναι απαραίτητα να διαθέτουν οι εργαζόμενοι, ποια είναι τα εμπόδια, τα εμπόδια δηλαδή που εμποδίζουν τις επενδύσεις σε παλαιές βιομηχανικές περιοχές και θα ήθελα επίσης να εξετάσω ποια εργαλεία είναι διαθέσιμα για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση. Ποιες δηλαδή χρηματοδοτικές αναγκαιότητες και ποιες χρηματοδοτικές δυνατότητες προσφέρουν τα ταμεία. Μετά από αυτό να εξεταστεί ποιες είναι οι επιπτώσεις για τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιες διασυνδέσεις υπάρχουν με την αστική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική και εδώ θέλω να τα μελετήσω αυτά και στην βάση παραδειγμάτων, γιατί σωστό είναι να γίνει σε μεγάλη έκταση. Έχουμε λάβει, για παράδειγμα, το Μάντσεστερ, την Λίλη και την Λιέγη. Παλαιές, δηλαδή, περιοχές εξόριξης άνθρακα και χαλιβουργίας. Όπως σε αυτές βασίστηκε βέβαια η Ένωση της Ευρώπης αρχικά και να εξεύρουμε κάποια εργαλεία τα οποία πρέπει να αναπτυχθούν για να στηρίξουν την ανάπτυξη αυτών των περιοχών που πλήττονται από τις διαφθορτικές αλλαγές και που έχουν περάσει μια ιστορία οι περιοχές αυτές πότε καλύτερα πότε χειρότερα. Αυτός είναι ο στόχος της έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας και θα χαρώ ιδιαίτερα εάν λάβω υποστήριξη από τις και τους συναδέλφους και βέβαια και προτάσεις και παρατηρήσεις. Thank you very much Is there any question? Ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις. Όχι. Τότε κλείνεται η συνεδρίασή μας. Καλό σας βράδυ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου. Γεια σας.